Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, όπω ξέρετε έχει λάβει χώρα ένα τρομερό σεισμό στο Νεπάλ. Ο αριθμό των θυμάτων έχει